Έτσι Κοπεχάγη έδειξε ότι θα κερδίζαμε 33 δι και εκείνη 18 δι από με τέτοια ρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Κέλλη, συνελήφθησαν όλοι οι οφθαλμοί και μπορώ να δώσω το λόγο στον Επίτροπο